ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ σημαντική ψηφοφορία. Καθίστε παρακαλώ. Colleagues, please take your seats. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, na początek chciałem Państwa poinformować. Θέλω να σας πληροφορήσω καταρχήν κυρίες και κύριοι